σε διάταξη. ευχαριστώ. Περνάμε λοιπόν ε, στην πρώτη ψηφορία για την έκθεση Φεράρα, απλή ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Άρχεται ψηφοφορία. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία. Συγχαρητήρια κυρία Φεράρα. Έχουμε και άλλη δικιά σας έκθεση. Μείωση της... Ε, όχι, πρόκειται για την εκτροπή των βασικών φαρμακευτικών προϊόντων. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Και αυτή η έκθεση εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία. Συγχαρητήρια κυρία εισηγήτρια. Έκθεση Βιέγκας Ψηφοφορίες σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του πριγκιπάτου της Ανδόρας για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Και εδώ συντριπτική πλειοψηφία, συγχαρητήρια ε, συνάδελφε Βιέγκα. Έκθεση Γκουαλτιέρη, διορισμό νέου εκτελεστικού διευθυντή τη Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. Πρόκειται για απλή ε, μυστική ψηφοφορία. Θα δείτε λοιπόν ότι το λαμπάκι θα είναι μπλε, ανεξάρτητα με το τι θα ψηφίσετε. Ψηφίζουμε παρακαλώ. η ψηφοφορία. Εγκρίνεται η έκθεση. Πάμε στην έκθεση της συναδέλφου Κινίτσι για τις δικονομικές εγγύησεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Ε, ψηφίζουμε παρακαλώ. Είναι 78 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Καταπίπτει το ένα. Ψηφίζουμε τώρα για την πρόταση της Κομισιόν στο σύνολό της υπέρ κατά αποχές. <clears throat> Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στο νομοθετικό ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Ε, συγχαρητήρια κυρία Κινίτσι. Ε, συνάδελφος Γκάια υπέβαλε μια έκθεση για τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2017, ε, τμήμα 3. Ψηφίζουμε καταρχήν για την τροπολογία υπερθυμών 25, υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 26, ονομαστική ψηφορία, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Τροπολογία υπαριθμών 5. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πάμε στην τροπολογία 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επίσης απορρίπτεται. Τροπολογία 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 29. Ονομαστική ψηφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Abstimmung geschlossen. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε η τροπολογία 30. Πάλι με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Και αυτό απορρίπτεται. Η τροπολογία 8 ε, της ομάδας EFTD. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται και ψηφίζουμε ε, για την 31 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Πάμε στην τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 32 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα ονομαστική ψηφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Και έτσι λοιπόν ε, ψηφίζουμε τώρα για την τροπολογία 10. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 33 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 11 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 21 υπέρ κατά αποχές ε, πρέπει να το επαληθεύσουμε παρακαλώ για την 21 ηλεκτρονική επαλήθευση. Έκλειση ψηφοφορία εγκρίνεται. Έτσι λοιπόν ε, το αρχικό κείμενο καταπίπτει. Πάμε στην ε, τροπολογία 34. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η τροπολογία 35, ονομαστική ψηφοφορία, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Και αυτή και Πάμε στη 12. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Πάμε στην 36. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Πάμε στην 37. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 38 ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε ψηφοφορία. Απορρίφθηκε επίσης. Πάμε στην τροπολογία υπαριθμών 1 των πρασίνων. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Ε, λυπάμαι. Πρέπει να κάνουμε ένα προβούμε σε παλήθευση. Παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Η 13. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 15. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. απορρίπτεται. Η 16, πάλι μονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Και αυτή απορρίπτηκε. Η 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 17 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται η 22 ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία υπαριθμών 40 και πάλι με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. απορρίπτεται η 41 σε δύο τμήματα ε, και τα δύο μονομαστική ψηφοφορία. Πρώτα για το πρώτο. Ε, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίθηκε ξεκάθαρα. Πάμε στο δεύτερο τμήμα. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 23 των Σοσιαλδημοκρατών, πάλι με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε για την 42, επίση ε, με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. απορρίπτεται. Η 18 του, της πολιτικής ομάδας EFTD, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 19. Πάλι ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. απορρίπτεται. Η 43 ε, χειρός υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 44 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 2 των πρασίνων ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε για την υπαριθμόν 4, επίσης ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Πάμε στην τροπολογία υπαριθμών 3 ε, και πάλι ονομαστική ψηφοφορία. Έκλειση ψηφοφορία. και αυτή απορρίφθηκε. Τροπολογία υπερθυμών 6 διανατάσεως της χειρός. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 24 της ενωμένη αριστερά σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Άρα καταπίπτει το δεύτερο τμήμα και ψηφίζουμε συνολικά για το ψήφισμα ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. έκλεισε η ψηφοφορία. Γκρίθηκε το ψήφισμα. Συγχαρητήρια κύριε Γκάια. Πάμε τώρα στην έκθεση της συναντέλφου Χούμπνερ που αφορά στη διοργανική συμφωνία για την βελτίωση της νομοθεσίας. Η τροπολογία υπερθμονένα υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, για το 2 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για τη 2 του αρχικού κειμένου. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 7 αρχικό κείμενο, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία, ψηφίζουμε παρακαλώ. εκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η 4 της πολιτικής ομάδας, η FTD, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η δύο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η έξι υπέρ κατά αποχές Επίσης απορρίπτεται αρχικό κείμενο της παραγράφου 12 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 8 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Και ψηφίζουμε συνολικά για το ψήφισμα ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Κλείσε η ψηφοφορία. εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία. Συγχαρητήρια κυρία Χύπνα. Και πάμε τώρα σε διάφορες προτάσεις ε, ψηφίσματος για τη συμφωνία για τον καπνό συμφωνία PMI. Το πρώτο είναι πρώτες ψηφίσματος της Ενωμένης Αριστεράς. Ψηφίζουμε ε, για την δύο αρχικό κείμενο, ένα ε, περ κατά αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα, παράγραφος 5 του αρχικού κειμένου σε δύο τμήματα, ονομαστική ψηφορία. Για το ένα ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, επίσης με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Πάμε στην τροπολογία υπεριθμών 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 1. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Κατόπιν τούτου πάμε στη 2. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Η ίδια πλειοψηφία. Αν θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση, εντάξει, ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την υπαριθμόν 2. Έκλεισε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Ε, πάμε τώρα στο αρχικό κείμενο του ψηφίσματος, παράγραφος 8, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ονομαστική ψηφοφορία για την 10 του αρχικού κειμένου. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, λυπάμαι ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε για την 3 παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Πάμε ε, σε ονομαστική ψηφοφορία για το αρχικό κείμενο του 12. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Του 11, με συγχωρείτε, του 11. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Και πάμε στο αρχικό κείμενο 12, ε, ονομαστική ψηφοφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία. και αυτό απορρίπτεται. Πάμε στην τροπολογία υπερθμών 4. Υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση. Λοιπόν, ηλεκτρονική επαλήθευση για την 4. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Πάμε στην 5. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Γκρίνεται. Πάμε στην 6. Διανατάσεις της χειρός. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτή. Και ψηφίζουμε για το ψήφισμα στο σύνολό του. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται και κατόπιν τούτου αφού απορρίφθηκε ε, το πρώτο σχέδιο πάμε στην κοινή πρόταση τριών πολιτικών ομάδων Πρασίνων, EFDD και Χριστιανών Δημοκρατών ψηφίζουμε για το πρώτο τμήμα υπέρ παρακαλώ του 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα του 3 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται μισό λεπτό ηλεκτρονική επαλήθευση επαλήθευση του δεύτερου τμήματος έκλειση ψηφοφορία εγκρίνεται εγκρίθηκε παράγραφος 4 του αρχικού κειμένου υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία υπαριθμών 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Για την 1 παρακαλώ ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Η 11. Αρχικό κείμενο, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 3. Ονομαστική ψηφοφορία. Η... Μισό λεπτό. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πάμε στην ονομαστική ψηφοφορία για το αρχικό κείμενο της παραγράφου 14. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίθηκε και ψηφίζουμε τώρα για το ψήφισμα στο σύνολό του υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές Νομίζω ότι καλύτερα να προβούμε σε επαλήθευση όσον αφορά την κοινή πρόταση ψηφίσματος. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία, η επαλήθευση. Εγκρίθηκε με σαφήνεια αυτή η πρόταση ψηφίσματος ως εκ τούτου, ως εκ τούτου λοιπόν καταπίπτουν οι, οι υπόλοιπε ψηφοφορίες και καταπίπτουν τα υπόλοιπα ψηφίσματα και έκλεισε η ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι.